Καθίστε παρακαλώ. Για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Θα ήθελα καταρχήν να εξετάσουμε το σχέδιο μερίσης διάταξης. Μήπως έχετε παρατηρήσεις για το σχέδιο. Όχι, οπότε θα τηρήσουμε το σχέδιο μερίσης διάταξης. Έχετε λάβει και τα πρακτικά της συνεδρίασης της Δευτέρας Δεκεμβρίου και αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, αύριο δηλαδή, θα θεωρήσουμε ως συγκεκριμένα τα πρακτικά. Έχω κάποιες ανακοινώσεις. πριν περάσουμε στην κυρίως ημερήσια διάταξη. Η έκθεση Βανίστερ Ρόι για την πράσινη βίβλο με θέμα το μέλλον της πολιτικής συνοχής έχει προκαλέσει σωρία τροπολογιών, γι' αυτό και ο κύριος Βανίστερ Ρόι ζήτησε μία παράταση του χρόνου προκειμένου να συγκροτήσει κάποιες συμβαστικές λύσεις. Γι' αυτό και η ψηφοφορία της έκθεσης Βανίστερ Ρόι αναβάλλεται για την επόμενη μας συνεδρίαση του Φεβρουαρίου. Μετά από διαβούλευση με συντονιστές των πολιτικών ομάδων, συμφώνησα και εγώ να υποστηρίξει η Επιτροπή μας μία προφορική ερώτηση μετασυζητήσεως με θέμα το σχέδιο δράσεως της κινητικότητας της πόλης που είχε εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά καθυστερεί η εφαρμογή του. Είχε γίνει σχετική συζήτηση στο Στρασβούργο την προηγούμενη Δευτέρα και εκεί μας εκπροσώπησε ο κύριος Ποπή που παρακολουθεί, όπως ξέρετε, εκ του σύνεγγης ε, τη δρομολόγηση αυτού του σχεδίου. Και έγινε από κοινού συζήτηση με την Επιτροπή Μεταφορών. Έχω να σας υποβάλω και κάποιες προτάσεις των συντονιστών για ορισμό εισηγητών. Σε ό,τι αφορά την έκθεση για το Γενικό Κανονισμό των Ταμείων, οι σοσιαλιστές προτείνουν την κυρία Γκαρθία Πέρες για την έκθεση που αφορά τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτείνει τον κύριο Αγγελάκα για τη γνωμοδότηση που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Απασχόλησης με θέμα τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι σοσιαλιστές προτείνουν την κυρία Μαδέιρα και για την γνωμοδότηση που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με θέμα το σχέδιο ανάκαμψης προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι σοσιαλιστές προτείνουν τον κύριο Κυρίλοφ. Μπορούμε να εγκρίνουμε τις προτάσεις αυτές για, για τον ορισμό των εισηγητών που έκαναν οι συντονιστές μας. Πολύ ωραία. Θα ήθελα πλέον να ενημερώσω ότι ο συνάδελφός μας, ε, Φιλίπ Πέτρου, εξελέγει στην Ρουμανική Βουλή και τον συγχαίρομαι θερμά για την εκλογή του. Θα αντικατασταθεί λοιπόν στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή από τον κύριο Αλεξάνδρου Νάζαρη. Υπάρχει όμως ένα τυπικό πρόβλημα εδώ. Στη γνωμοδότηση που είχε αναλάβει ο κύριος Φιλίπ ε, την εκπόνησε και θα ψηφίσουμε αύριο να έχει προβλεφθεί η ψηφοφορία στην αυριανή συνεδρίαση. Όπως ξέρετε δεν μπορούμε να υποβάλουμε στην Ολομέλεια μια έκθεση γνωμοδότηση ε, κάποιου που δεν είναι πια ευρωβουλευτής. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από το ΕΛΚ να μας ε, επισημάνει ποιος θα αναλάβει την έκθεση. Ο κύριος Ναζάρο, ο αναπληρωτής, ο βουλευτής που θα λάβει τη θέση του κυρίου Πέτρου ή ο κύριος Βανίστερ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, το στη Γερουσία την ε, Ρουμανική έχει εκλεγεί και γι' αυτό ακριβώς από, θα, θα γίνει το αντίθετο τώρα. Ναι. Eh, ο συντονιστής ακριβώς θα περάσει, ναι, το σημειώνουμε αυτό. Θα προχωρήσουμε. Έτσι ακριβώς ε, όπως ε, προβλέπει ο κανονισμός μας. Για το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης θα ήθελα ένθερμα να καλωσορίσω τον κύριο Κούνεκ, Τσούνεκ, Τσούνεκ, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Τσεχίας και υπουργό περιφερειακής ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ο οποίος και θα μας αναλύσει τις προτεραιότητες της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Χιούμπνερ, την Επίτροπό μας, Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που όπως προβλέπετε σήμερα το απόγευμα θα μας παρουσιάσει τις τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την κοινοβουλευτική μας δουλειά με την χρήση των κονδυλίων και του Ταμείου συνοχής. Ε, με, πριν λίγο από αυτές τις παρουσιάσεις θα ήθελα να σας κάτι. ότι θα έχουμε μία μετάδοση αυτής της συνομιλίας και αυτών των παρουσιάσεων μέσω του συστήματος που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι θα έχουμε μια απευθείας ε, πρόσβαση όλων των πολιτών μέσω του ίντερνετ. Ε, χαίρομαι για αυτό που γίνεται, για το γεγονός αυτό. Πιστεύω ακριβώς ότι για τα μέλη της Επιτροπής μας είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό να είναι σχεδόν η πρώτη, η πρώτη κοινοβουλευτική επιτροπή που πειραματιζόμαστε με τον ε, τρόπο αυτό μετάδοσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πώς ε, μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με τον κύριο Τσούνεκ και για την κυρία Χίμνερ, θα ήθελα κάτι να σας πω, σίγουρα θα το έχετε πληροφορηθεί διότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή τη ζητούν την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έτσι να εγκρίνουμε τάχιστα τα μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος του οικονομικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι Όλα αυτά που έχουν σχέση με την κοινοφτευλική μας εργασία, τα διαφορετικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και τα κονδύλια να μπορέσουν ε, να καταλήξουν όσο γίνεται συντομότερα στα κράτη-μέλη, να υπάρξει ρευστότητα, ρευστό στην αγορά και έτσι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. για τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων ε, σήμερα το απόγευμα σε μια έκτακτη συνάντηση που έχω συγκαλέσει στο τέλος αυτής της συνεδρίασης ε, ο στόχος έλεγα και που ανακοινώθηκε στους εισηγητές ε, και πριν από λίγο το εγκρίναμε Ο στόχος είναι σε μια έκτακτη συνάντηση της κοινοβουλευτική μας Επιτροπής να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τις 9 Μαρτίου. 9 Μαρτίου και έτσι η διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών να μπορέσουν να αποφασίσουν να το συμπεριλάβουν στην Ολομέλεια αν γίνεται το τέλη Μαρτίου διαφορετικά έτσι και αλλιώς μία από τις δύο Ολομέλειες συνόδους όπως έχουν προβλεφθεί του Απριλίου την Σύνοδο. Στη συνάντηση αυτή των συντονιστών ε, θα δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε την ε, διαδικασία αυτή και θα ήθελα να τονίσω χωρίς ε, να παραβούμε τα όσα έχουμε σαν δυνατότητες στην όλη νομοθετική διαδικασία και θα μπορούσαμε αύριο να επανέλθουμε στο θέμα αυτό μετά από όσα ε, συζητούν, θα συζητηθούν στην συνάντηση των συντονιστών και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Τσούνεκ, ε, τον ε, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Δημοκρατίας Τσεχίας, να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Τσεχικής Προεδρίας και τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι βουλευτές, καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ σήμερα να μιλήσω μαζί σας και να παρουσιάσω σε γενικές γραμμές την προσέγγιση της ε, Τσεχικής Προεδρίας προς την πολιτική συνοχής. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσω για δύο πράγματα. Σήμερα πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφέρω τις προτεραιότητες της ε, Τσεχικής Προεδρίας και κατόπιν να εξηγήσω τους στόχους μας όσον αφορά την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων για την αλλαγή του κανονισμού της ε, πολιτικής συνοχής. Μαζί με την Γαλλία και την Σουηδία η Τσεχία έχει ένα κοινό πρόγραμμα 18 μηνών και με βάση αυτό ορίστηκαν οι προτεραιότητές μας, οι οποίες είναι ε, τρεις, τρίπλες θα λέγαμε. Πρώτα απ' όλα αφορά την ε, συζήτηση που θα γίνει για την πολιτική συνοχής ε, μέχρι και τον Ιούνιο και αναμένουμε βεβαίως αυτά τα οποία θα πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης ε, σκοπεύουμε να παίξουμε ενεργό ρόλο στην ομαλή εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Και επίσης θέλουμε να συνεισφέρουμε στην επιτυχή οριστικοποίηση προγραμμάτων για το και κλείσιμο των προγραμμάτων για την περίοδο 2002-2006. Ε, θέλουμε επίσης να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος να μοιραζόμαστε τις ε, πληροφορίες ε, για να μπορέσουμε έτσι να απλοποιήσουμε την όλη διαδικασία εφαρμογής. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να συνεχιστεί η δημόσια διαβούλευση για την πολιτική εδαφική συνοχής. Μια διαβούλευση η οποία έχει ήδη και θα ήθελα εδώ πέρα να επισημάνω το ενδιαφέρον έργο το οποίο έχει επιτελεστεί στο Συμβούλιο επί Τσεχικής Προεδρίας είναι μια κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να συνεχίσουμε, να συνεισφέρουμε και εμείς στην συζήτηση αυτή που θα βοηθήσει τα θεσμικά όργανα και τους λοιπούς εταίρους ε, να έχουν μεγαλύτερη κατανόηση. Τέλος, ως Προεδρία θα παραμένουμε προσιλωμένοι σε αυτά τα οποία προκύπτουν από την χάρτα της λειψίας και την ε, εδαφική ατζέντα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και αυτά τα οποία αποφασίστηκαν και στα Συμβούλια Υπουργών και στο τελευταίο Συμβούλιο στην Μασαλία. Όσον αφορά λοιπόν το σχετικό ε, σχέδιο δράσης θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί, δηλαδή οι σχέσεις ανάμεσα στις πόλεις και την Ήπεθρο και παρά το ότι δεν σκοπεύουμε να αφιερώσουμε ένα συμβούλιο ειδικά στις πόλεις θα θέλαμε παρόλα αυτά να δοθεί κάποια προσοχή στην χάρτα της λειψίας και να δώσουμε βάρος ε, στις ε, βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πόλεων. Θα επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτές τις ε, δραστηριότητες, ε, σε πολλές επίσημες και άτυπες διασκέψεις που θα διοργανωθούν κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρία μα. Εδώ πέρα θα ήθελα να φερθώ συγκεκριμένα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Αρμοδίων για την ε, Περιφερειακή Πολιτική που θα οργανωθεί 23 και 24 Απριλίου στη Μαριάν Σκαλάσνια. Έχω ήδη λάβει επιβεβαίωση από την κυρία Ντανούτα Χιούμπνερ, η οποία θα είναι παρούσα και στις δύο ημέρες του ατύπου συμβουλίου θα παρουσιάσει τις θέσεις της ε, Κομισιόν καθώς και τα αποτελέσματα της διαβούλευσης επί της Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή. Η δεύτερη σημαντική εκδήλωση θα είναι ένα διεθνές συνέδριο για το, διεθνής διάσκεψη για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής που θα είναι στις 26-27 Μαρτίου στην Πράγα. Επιπλέον διάφορα θεσμικά όργανα θα διοργανώσουν ε, διάφορες διασκέψεις, π.χ. η Επιτροπή των Περιφερειών θα διοργανώσει αρχές Μαρτίου την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής ε, Πόλεων και Περιφερειών της ε, Ευρώπης στην Πράγα και θα έχουμε τον Φεβρουάριο την Ευρωπαϊκή ημέρα των πόλεων επίσης. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για το νομοθετικό μας πρόγραμμα. η σοβαρή αυτή οικονομική και δημοσιονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιες νομοθετικές προτάσεις. Η Προεδρία μας δεν θα αυστεί προσπαθειών για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σεβόμενη βεβαίως τις ευθύνες που έχουμε και ελπίζω εδώ πέρα να μας βοηθήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και οι πολίτες μας δεν θα ανεχτούν οποιαδήποτε καθυστέρηση. Τον ε, Νοέμβρη που μας πέρασε η Κομισιόν παρουσίασε τρεις σημαντικές νομοθετικές προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης. Αυτά τα πράγματα πρέπει να θεωρηθούν ότι συνδέονται, αποτελούν ένα τμήμα ενός ενιαίου πακέτου και έτσι τα αντιμετώπισε και το Συμβούλιο. Στόχος όλων αυτών των προτάσεων είναι να απλοποιηθεί η υπάρχουσα οδηγία για τα διαρθρωτικά μέτρα και να γίνεται, ε, να γίνει η ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Έτσι θα δοθούν κίνητρα και στην Ένωση και στα κράτη-μέλη <clears throat> για να εκταμιεύουν καλύτερα και γρηγορότερα τα σχετικά κονδύλια. Στα δε συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης και 12ης Δεκεμβρίου 2008 αναφέρεται πως ε, καλεί το Κοινοβούλιο, Κομισιόν και Συμβούλιο να αναλάβουν τα σχετικά μέτρα, το, να λάβουν τα σχετικά μέτρα το τσομότερο δυνατόν, σεβόμενοι τις δημοσιονομικές προοπτικές και τις διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται στην Διαθεσμική Συμφωνία. Και όλα αυτά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Το Συμβούλιο αντέδρασε γρήγορα σε αυτή την ε, έκκληση. Μπορώ να πω ότι ελαχιστοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις παρά το ότι αρκετά κρατημέλη είχαν αντίθετη άποψη και τελικά όλες οι αλλαγές σε οποίες παρουσίασε το Συμβούλιο εγκρίθηκαν από την Κομισιόν οπότε σήμερα μπορώ να κάνω αρκετές ανακοινώσεις ότι πρώτα απ' όλα το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να τροποποιήσει τον κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να επεκτείνει τα είδη δαπανών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από αυτό το Ταμείο. Να τονίσω πως ε, το Συμβούλιο δεν έχει επιβάλει κάποιες ε, Αλλαγέ. Η Κομισιόν δεν έχει επιβάλει κάποιες αλλαγές και ελπίζουμε το ίδιο θα κάνει και το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε μια γρήγορη συμφωνία για το τελευταίο μέρος των αλλαγών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά τις επενδύσεις ε, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις απές τομέα της στέγασης. Τέλος, συμφωνούμε με την Κομισιόν πως οι επενδύσεις όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες είναι πολύ σημαντικές, ειδικά σε αυτή την κατάσταση κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει ελλείψεις φυσικού αερίου. Πρέπει να επενδύσουμε σε μόνωση κτηρίων, σπιτιών που μπορούν να μας οδηγήσουν σε πολύ μεγάλες οικονομίες ενέργειας. Να τονίσω πως αυτό είναι το πιο πολύπλοκο μέρος της συζήτησης μεταξύ των κρατών μελών. Τα περισσότερα κράτη-μέλη συμφωνούν με τις επενδύσεις στην στέγη όπως προτείνει η Κομισιόν, αλλά κάποια κράτη-μέλη δεν υποστηρίζουν την επιλεξιμότητα από τα διαρθρωτικά ταμεία αυτών των δαπανών και ως συμβαστική λύση αποφασίστηκε να εισαχθεί ένα κατόφλι 4% των συνολικών ευρωπαϊκών δαπανών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τέλος, να σας πω γιατί αλλάξαμε τον ορισμό των εισοδημάτων των με νοικοκυριών χαμηλών εισοδημάτων για την πολιτική κοινωνική συνοχή. Όπως ξέρετε δεν υπάρχει ε, ε, ευρωπαϊκός ε, ορισμός της κοινωνικής στέγης λόγω των διαφορετικών καταστάσεων που επικρατούν. Οπότε θεωρήθηκε πως ο ορισμός που θα κρίνει την επιλεξιμότητα θα είναι αρμόδια των κρατών μελών. Τρίτον, και η Προεδρία γνωρίζει τις προηγούμενες εκθέσεις που είχε εθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα ιδιαίτερα την έκθεση του κ. Αντριάν που υιοθετήθηκε την άνοιξη του 2007. Θεωρώ πως οι αλλαγές που προτείνονται από το Συμβούλιο θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου γιατί έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια όσον αφορά την κοινωνική στέγη, την πολιτική στέγαση. Τώρα όσον αφορά τους ε, προσπάθεια να υπάρξουν μέγιστοι κοινοί κανόνες σε όλα τα ταμεία, η Προεδρία και η Κομισιόν πρότειναν ε, μέτρα για τα καταποκοπήν ποσά όπως πρότεινε η Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η ε, ημερομηνία είναι η 1η Αυγούστου 2006 με αναδρομική ισχύ βεβαίως. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στον τελευταίο κανονισμό, στον κανονισμό πολιτικής συνοχής. Το Συμβούλιο θα ζητήσει από το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει με την τροποποίηση κάποιων την διαχείριση του ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Ε, εμείς αποδεχόμαστε την πρόταση αυτή με κάποιες ε, αλλαγές τεχνικής φύσης, οπότε θα ήθελα να τονίσω την πιο σημαντική πτυχή, δηλαδή την αύξηση των προκαταβολών την ε, παροχή άρα προκαταβολών και το 2009 για τα νέα κρατημέλη με αύξηση από το 2% στο 4% και όσον αφορά τα παλαιότερα κρατημέλη θα έχουμε μια νέα πληρωμή που δεν υπήρχε στο παρελθόν και ανέρχεται σε 2,7% κοινοτική συνεισφορά για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτές οι προκαταβολές θα καταβληθούν το των δυνατόν έτσι ώστε οι φορείς διαχείρισης να μπορούν να ξεκινήσουν τα νέα έργα ώστε να δυνατόν γρηγορότερα με στόχο να επιταχυνθούν οι πληρωμές και η εφαρμογή προγραμμάτων πολιτικής συνοχής. Θεωρώ πως θα συμφωνήσει και το Κοινοβούλιο με το Συμβουλίο και την Κομισιόν και θα μπορέσουμε να δράσουμε γρήγορα. Γιατί η γρήγορη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτές τις νομοθετικές προτάσεις αποτελεί και την δική μας προτεραιότητα όσον αφορά το νομοθετικό μας πρόγραμμα. Έθελα τώρα να εκφράσω και τις προσωπικές μου ευχαριστίες στην ε, Γαλλική Προεδρία η οποία αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου, όσον αφορά τις ε, συζητήσεις για συμβιβαστικά κείμενα στο Συμβούλιο. Ήθελα να τονίσω την σημασία επίσης και της ε, βοήθειας από την Κομισιόν, γιατί ακολουθούμε ένα κοινό στόχο να καταλήξουμε πολύ γρήγορα σε μια συμφωνία για τις τρεις αυτές προτάσεις που ανέφερα και θεωρώ πως η Κομισιόν μπορεί να υποστηρίξει τα αποτελέσματα τα οποία επέτυχε το Συμβούλιο και νομίζω αυτό μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να συνοψίσω με αρκετά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Τώρα εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να ευθύσει γρήγορα μια γνωμοδότηση για αυτές τις νομοθετικές προτάσεις. Εμείς ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει εγκαίρος έτσι ώστε να υιοθετήσουμε αυτούς τους κανονισμούς χωρίς ε, καθυστερήσεις. Η Προεδρία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμες και ανοιχτές να δουν όλες σας τις τροπολογίες, να συζητήσουν όλες τις τροπολογίες και θα ήθελα τελειώντας να πω το εξής. Ε, ίσως γνωρίζετε πως αποφάσισα να αποχωρήσω από την κυβέρνηση της χώρας, της ε, Τσεχίας και θέλω να σας διαβεβαιώσω πως ε, θα υπάρχει συνέχεια και διαδοχή χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Φόμποντα, τον οποίο πρότεινα εγώ στον ε, Πρωθυπουργό, θα συνεχίσει το έργο αυτό όμαλα, οπότε σας διαβεβαιώ πως ο ανασχηματισμός αυτός δεν θα επηρεάσει την ποιότητα του έργου μας. Ευχαριστώ. Σίγουρα αυτό και θα συμβεί. Σας προτείνω τώρα το λόγο να λάβει η κυρία Επίτροπος, κυρία Χίμπνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριε Αντιπρόεδρε τη Τσεχική Κυβέρνηση, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερω που μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου ξαναβρίσκομαι στην Επιτροπή σα και σα εύχομαι καταρχήν καλή χρονιά, πολλέ επιτυχίε και να ευχαριστήσω θερμά τον Αντιπρόεδρο Τσούνεκ για την παρουσίασή του αλλά και για τις δεσμεύσεις της Τσεχικής Προεδρίας ε, ε, και την προσήλωσή της στην πρόοδο σε ό,τι αφορά βασικά τομεί πολιτική και στη διάρκεια τη τυχική προεδρία και ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σα σε ό,τι αφορά την πρόθεση των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση του κανονισμού για την πολιτική συνοχή. Δράτω με τι παρούσε ευκαιρίε για να σα δώσω κάποιε σύντομε πληροφορίε για κέρια ζητήματα που βρίσκονται στο πρόγραμμα εργασιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική συνοχή αλλά και ε, σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις στον κανονισμό. Όπως ξέρετε, βρισκόμαστε τώρα στη φάση της έναρξης ε, των αγενείων της νέας δημοσιονομικής περίοδου 2007-2013 και προσπαθούμε να, ε, να εγκρίνουμε και την, ε, τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης που είναι σημαντικό τμήμα της διαδικασίας διαχείρισης της πολιτικής συνοχής. Μέχρι στιγμής έχουμε λάβει τα δύο τρίτα για το Περιφερειακό Ταμείο από, το, από τις συνολικές αξιολογήσεις συμμόρφωσης που καλύπτουν 80 περίπου 100 των πληρωμών. Και ευελπιστώ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα λάβουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία ε, της διαχείρισης ώστε να βεβαιωθούμε για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλές εκκλήσεις ε, για τρέχοντα προγράμματα από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και επιμένουμε σε όλες μας τις ε, συναντήσεις, ε, επιμένουμε στα ποιοτικά προγράμματα. Κάτι που φυσικά απαιτεί και μια υγιή δημοσιονομική διαχείριση. Και μάλιστα η αξιολόγηση της συμμόρφωσης είναι ένα νέο εργαλείο που μας διαβεβαιώνει για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των ταμείων γενικά και του συγκεκριμένου ταμείου ιδιαίτερα. Ολοκληρώνουμε επίσης και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από ένα χρόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής. Και αύριο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα γίνει συζήτηση και ακρόαση για την απαλλαγή για το 2007. Σε ό,τι αφορά το αριθμό απορρόφησης ε, των περσινών ε, κονδυλίων των ταμείων, στα τέλη του μήνα θα μπορέσω να σας ε, δώσω πιο διεξοδικά και ακριβή στοιχεία για το βαθμό απορρόφησης. Μέχρι στιγμής πάντως υπερβαίνουμε κατά κανόνα το 90% ε, κατά μέσο όρο για όλα τα διαφορετικά ταμεία και τα κράτη-μέλη και περίπου τα μισά κράτη-μέλη έχουν ε, κατορθώσει βαθμό απορρόφησης το 95% των δαπανών μέχρι τα τέλη του προηγούμενου έτους. Και μάλιστα γίνεται τώρα μια παράταση της περίοδου επιλεξιμότητας, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κατά τη γνώμη μου για την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων στα περισσότερα για να μην πω σε όλα τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, ε, συνεχίζουμε τη διαδικασία θέση των θεμελίων για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής και μετά το 2013 και μάλιστα έχουμε δημοσιεύσει τα αποτελέσματα αξιολόγησης της περίοδου 2000-2006 και το αναφέρω στα πλαίσια της συζήτησης για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής γιατί από την αξιολόγηση της προηγούμενης περίοδου θα αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα και για την προετοιμασία της μελλοντικής πολιτικής. Κάτι που βοηθάει στη συζήτηση για το μέλλον της ε, πολιτικής μετά το 2013 είναι η πρόσφατη δημοσίευση της έκθεσης της Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης για την περίοδο μέχρι το 2020 με ανάλυση των συνεπειών των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες μέχρι το 2020 και φαίνονται τα ευαίσθητα σημεία των περιφερειών σε διαφορά τις κλιματικές αλλαγές, τις δημογραφικές αλλαγές, τις πιέσεις λόγω της παγκοσμιοποίησης, το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Θα εξεταστούν υπό το πρίσμα όλων αυτών των προκλήσεων ε, τα προβλήματα των ε, ευρωπαϊκών περιφερειών για να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε και τις δικές μας προτεραιότητες ανάλογα με τα συμπεράσματα αυτά. Μάλιστα, πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που αναμένεται προς τα τέλη Μαρτίου για την πολιτική αυτή και ευελπιστώ ότι τον Απρίλιο θα μπορέσω ήδη να δημοσιεύσω τους προσανατολισμούς, τους μελλοντικούς προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής ε, Πολιτικής Συνοχής. Κάτι που θα συζητήσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα γίνει στο Μπάτ, Μαριάνς και Λάζνιε, τον Απρίλιο. Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζονται οι δημόσιες διαβουλεύσεις για την εδαφική ε, συνοχή και αναμένεται η πράσινη βήλωση στα τέλη Φεβρουαρίου και τα κατακτικά σχόλια για τη διαδικασία διαβούλευσης που θα σας υποβάλω στην Πράγα στις αρχές του Μαρτίου στη διάσκεψη κορυφής ε, των Ευρωπαϊκών Πόλεων που οργανώνει η Επιτροπή των Περιφερειών. Επίσης τον Ιούνιο θα υιοθετήσουμε την, έκτη έκθεση πρόοδου για την οικονομική κοινωνική συνοχή και θα γίνει και μια σύνοψη συζήτησης για την εδαφική συνοχή. Πάντως ε, το αναλυτικό τμήμα της έκθεσης ε, φέτος θα αφιερωθεί στη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε ε, περιφερειακό επίπεδο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι διανύουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Καινοτομίας και Δημιουργικότητας. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες προς την Τσεχική Προεδρία για την προσήλωση που δείχνει στη συζήτηση για την, ε, για την διάσταση πόλεων και υπαίθρου σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διαρθρωτικές δράσεις και ευελπιστούμε σε μια ε, επικοδομητική συζήτηση στη συνδιάσκεψη της Πράγας. Η Τσεχική Προεδρία έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει το πρώτο πρόγραμμα δράσης από, την, από το εδαφικό πρόγραμμα εργασιών με ύψιστη προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Στη διάρκεια της Τσεχικής Προεδρίας θα ολοκληρώσουμε και τη νέα μας προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Την στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας που θα υποβληθεί με τη μορφή ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ευθυνθεί κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη Μαΐου και θα υποβληθεί κατόπιν στο Συμβούλιο. Ελπίζω ότι θα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα νέο στοιχείο στην πολιτική συνοχή που εστιάζεται στα διασυνοριακά προγράμματα και ε, εντοπίζεται σε πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα περιφερειών που έχουν κοινά ιστορικά στοιχεία και κοινά στοιχεία ταυτότητας. Έχουμε, ε, ζητούμε για παράδειγμα από τις χώρες ε, γύρω από το Δούναβι να έχουν ε, παρόμοια προσέγγιση για την λεκάνη του Δούναβιου. Αυτό θα επηρεάσει και τη μελλοντική αρχιτεκτονική της ε, πολιτικής συνοχής και δαφικής συνεργασίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες και εργασίες μας και για τις υπεραπόμακρες περιοχές. Πέρυσι τον Οκτώβριο είχαμε δημοσιεύσει μία ανακοίνωση που μεταθέτει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις περιοχές αυτές και μεταφέρει την ε, έμφαση όχι μόνο στις αδυναμίες και τα προβλήματα αλλά και στα ε, γερά σημεία, στα δυνατά σημεία αυτών των περιοχών. Επίσης θα οργανώσουμε φέτος και το φόρουμ των υπεραπόμακρων περιοχών που ε, θα λάβει χώρα του χρόνου και δεν θυμάμαι σας το είχα πει άλλη φορά ένα άλλο τμήμα της, του σχεδίου εργασίας μας για φέτος είναι και η η ανακοίνωση για, για την πρώτη πενταετία του Ταμείου Αλληλεγγύης που στοχεύει στη βελτίωση φυσικά αυτού του εργαλείου. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ανάκαμψης που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου, θα ήθελα να σας πω το εξής. Συμφωνήσαμε να χρησιμοποιήσουμε, να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες ε, για την ε, εύρυθμη λειτουργία της πολιτικής συνοχής παρά την κρίση που σοβεί και να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες και τις περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης να επενδύσουν ε, τους πόρους της, ε, να επενδύσουν τους πόρους της πολιτικής συνοχής με τρόπο που να επιταχύνει την έξοδό μας από την οικονομική και δημοσιονομική κρίση. Πάντως όλοι οι συνάδελφοι της ε, Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης συνεργάζονται στενά με όλες τις αρμόδιες αρχές που διαχειρίζονται το προγράμμα ώστε να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το δυναμικό κάθε προγράμματος για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες και να, να επιταχυνθεί ο ρυθμός των επενδύσεων. Γιατί πιστεύουμε ότι στο ισχύον νομικό πλαίσιο Υπάρχει ελαστικότητα που μας επιτρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ήδη, χωρίς να περιμένουμε την αναθεώρηση του κανονισμού. Για παράδειγμα, οι διαχειριστές μπορούν να κατανείμουν το ε, ποσοστό κατανομής των διαφόρων ε, συμβολών στα προγράμματα, δίνοντας ήδη από την αρχή του προγράμματος το 100% του επιλέξιμου ε, κόστους της Ευρωπαϊκής Συνεισφοράς. ή κάνοντας μια διαφορετική κατανομή στη διάρκεια της περίοδου. Αυτή η ελαστικότητα προβλέπεται ήδη από την τρέχουσα νομοθεσία. Όπως είπε και ο Τσέχος Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι προς το συμφέρον μας να επιταχύνουμε τα πράγματα για να εξέλθουμε από την κρίση και αυτό θα γίνει χάρη στη συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων, ώστε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τις μεταρρυθμίσεις της τροπολογίας στον κανονισμό. Και μετά την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δευτέρας Δεκεμβρίου σας έθεσα ήδη τις προτινόμενες τροπολογίες για τον κανονισμό. Άλλωστε έχω ήδη συναντηθεί στο Στρασβούργο με τους συντονιστές, με τους εισηγητές συγγνώμη και τον ε, Επίτροπο Σπίτλα, καθώς και εκπρόσωπο της Τσεχικής Προεδρίας και μάλιστα ο Υπουργός Τσούνεκ ε, σας παρουσίασε μεγαλύτερες λεπτομέρειες ε, τη συμβαστική λύση που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο. Ίσως ε, δεν θα έπρεπε να το πω, αλλά το Συμβούλιο μας εξέπληξε πολύ ευχάριστα, γιατί με πολύ ταχύ ρυθμό δέχτηκε τις νέες τροπολογίες και ε, η Τσεχική Προεδρία εργάστηκε σε συνεργασία με την Γαλλική πολύ ε, σκληρά όλο το Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι τροπολογίες. Ελπίζουμε όλες αυτές οι νομοθετικές αλλαγές να συμπεριληφθούν στον κανονισμό, ώστε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ρευστότητα το συντομότερο δυνατό στις διάφορες περιφέρειες για τα προγράμματα και να μειώσουμε και το διοικητικό άχθος για να βελτιώσουμε την πρόσβαση ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα προγράμματα και να διευκολύνουμε τις διατυπώσεις για αυτές φυσικά με σεβασμό των δημοσιονομικών κανόνων και των κανόνων πρόσβασης στις ε, επενδύσεις, στις, στις συνεισφορές για τις επενδύσεις. Όλες αυτές τις τροπολογίες τις υπέβαλα εγώ το Δεκέμβριο και σας τις εξέθεσε και ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Τσούνεκ. Φυσικά όλες αυτές οι τροπολογίες έχουν διαφορετική αξία και σημασία για τους διαφόρους δικαιούχους της ευρωπαϊκής πολιτικής και σίγουρα επιπλέον ε, προκαταβολή θα είναι πολύ σημαντική αν και τα κράτη-μέλη δώσουν τη δυνατότητα κατανομής αυτής της ε, συμπληρωματικής προκαταβολής μεταξύ των δικαιούχων και να βοηθήσουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν τη ρευστότητά τους. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη προκειμένου να τα προετοιμάσουμε για να χρησιμοποιήσουν τις προτινόμενες τροπολογίες. Ήδη έγιναν οι πρώτες συνεδριάσεις με τα κράτη-μέλη γιατί σίγουρα άλλο η θεσμική προεργασία για την ε, έγκριση των τροπολογιών και άλλο η έμπρακτη εφαρμογή τους και η εξασφάλιση εφαρμογή τους από τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν αυτές τις νέες δυνατότητες όσο περισσότερο γίνεται. Είχαμε πολλές συζητήσεις και στις περιοχές. Επισκέφθηκα πρόσφατα πέντε περιοχές, περιφέρειες ε, και υπάρχουν τεράστιες προσδοκίες, υψηλότερες προσδοκίες και τεράστιες ανάγκες ε, από τις περιφέρειες. Γι' αυτό και βρήκαν μεγάλη απήχηση οι προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι προσβλέπουμε στη δική σας υποστήριξη. Θέλουμε να στηριχθούμε στην ε, μέχρι στιγμής πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί. Θέλουμε να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, όπως είπε και ο Χεράρτο Γκαλεότε, ώστε ήδη στο πρώτο τρίμηνο του έτους να εγκρίνουμε αυτές τις νομοθετικές ε, μεταρρυθμίσεις. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και εσάς και την Γαλλική Προεδρία για την τη ε, υιοθέτηση τροποποίησης του άρθρου 55 που ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για τις περιφέρειες και ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από τους δικαιούχους. Είναι, ήταν το πρώτο βήμα άλλωστε που κάναμε στο δρόμο της απλούστευσης. Τώρα έχουμε τις τελευταίες νομοθετικές προτάσεις, αλλά έχουμε ε, ήδη συγκροτήσει μια ομάδα εργασίας με, τα, με τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους των κρατών μελών, που προσπαθούν να απλουστεύσουν ακόμη περισσότερο την εφαρμογή της ε, πολιτικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ελέγχου και εποπτείας. Σε μια πλούστευση που δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής. Συμφωνώ πάντως με τον ε, Αντιπρόεδρο Τσούνεκ ότι ε, θα πρέπει να υποβληθεί και στα τέλη του Μαΐου και επίσης να έχουμε την παρουσίαση των πρώτων ε, αποτελεσμάτων της ομάδας αυτής της εργασίας και στη δική σας επιτροπή, αν σας ενδιαφέρει φυσικά, αν σας ενδιαφέρουν εργασίες αυτής της ομάδας. Πολλά είναι τα εκκρεμή θέματα και πολύ άριθμε αυτά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία θέτησης των τροπολογιών στον κανονισμό, με συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι πληροφορίες χρειάζεται και ό,τι υποστήριξη θέλετε από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε ώστε να κατανοήσετε πλήρως και τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και το περιεχόμενο των τροπολογιών. Ό,τι χρειάζεται ε, Είμαστε στη διάθεσή σας ε, για υλικό που ίσως θέλετε να, να μεταδώσετε στην πατρίδα σας, στην περιφέρειά σας. Είμαστε, επαναλαμβάνω, πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Προβλέπετε 35 λεπτών συζήτηση μέχρι τις 4.30. Παρακαλώ λοιπόν, επειδή αρκετοί έχουν ζητήσει το λόγο, να είστε σύντομοι στις παρατηρήσεις σας, περιληπτικοί όσον αφορά τις ερωτήσεις σας, επαναλαμβάνω, ώστε όλοι να λάβουν το λόγο. Και παρακαλώ, ένα πρώτο γύρο για τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και μετά έχουν ζητήσει πέντε το λόγο, πέντε συνάδελφοι και έτσι να κλείσουμε και τον κατάλογο των ομιλητών με αυτούς τους πέντε και να προχωρήσουμε σύμφωνα με αυτό. Από το ΕΛΚ ο συντονιστής ο κύριος Βανίστελ Ροή έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Εδώ πρόκειται για μία ειδική χρονιά, το γνωρίζετε. Εδώ εμείς ε, χρειαζόμαστε την υποστήριξη των πολιτών. Ε, θα είμαστε σε επαφή με τους πολίτες και για να ενισχύσουμε τόσα γίνονται εδώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και επί τόπου. Έχουμε ακόμα περίπου δύο μήνες για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το συγκεκριμένο. Γι' αυτό λοιπόν για μας είναι σημαντικό να έχουμε τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες από πλευράς Επιτροπής. Να τονίσω δύο-τρία πραγματάκια τώρα. Πριν από λίγο η Επίτροπος κυρία Χίμπνερ μίλησε για το recovery plan την ε, σχέδιο ανάκαμψης και μίλησε επίσης για απλοποίηση. Ναι, Πραγματικά αυτό που βρίσκεται μπροστά μας είναι ακόμα κάτι περισσότερο. Αναφέρεται μια ομάδα εργασία ε, που θα ασχοληθεί για τις διάφορες υπηρεσίες και για απλοποιήσεις και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν πριν από τις εκλογές για να πετύχουμε και ένα αποτέλεσμα. Η ερώτηση είναι εξή. Θα έχουμε νέες νομοθετικές ε, μεταβολές ε, κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής. Και για μας Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν γιατί διαπιστώσαμε ακόμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να έχουμε αλλαγές ας πούμε σε κάτι σε ένα κείμενο εδώ. Αυτό το ερωτώ στην Επίτροπο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της. Δεν είναι ότι έχει μόνο δύο-τρεις μήνες ζωής μπροστά της. Έτσι. Και επίσης αναφέρθηκε η ειδική κατάσταση για την οικονομική κρίση και για την βοήθεια που μπορεί να δώσει η Ευρώπη χάρη σε αυτά τα περιφερειακά ταμεία κλπ. Και τα κονδύλια. Λοιπόν, είναι ειδική στιγμή, γι' αυτό και χρειάζεται μια ειδική απάντηση. Δεν είναι τα συνηθισμένα πράγματα, δεν είναι business as usual, όπως τα πούμε στα αγγλικά, αλλά business as unusual. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Υπάρχει λοιπόν κάτι το επίγον, έτσι. Λοιπόν, και εμείς εδώ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενεργήσουμε τάχιστα και έτσι να λάβουμε αποφάσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα, να σεβαστούμε και τις προθεσμίες που έχουν τεθεί και έτσι πριν από τις εκλογές και μάλιστα πριν από το Μαρτίου αρχές Απριλίου να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και από τις διάφορες επαφές που είχα αναρωτιόταν όλοι πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε για να προσφέρουμε απτά αποτελέσματα, να τα δουν, να τα καταλάβουν οι πολίτες πριν ε, πάνε στις κάλπες. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να χάσουμε χρόνο. Και ακόμα κάτι, μίλησε η Επίτροπος για το Ταμείο Αλληλεγγύης οι προθέσεις ποιες ακριβώς είναι. Μπορείτε να μας πείτε και στο θέμα αυτό τι γίνεται, τι θέλετε ακόμα να συζητήσετε με το Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό και τι ακριβώς προσδοκεί η Επιτροπή σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης. Και ακόμη για τον Τσέχο Αντιπρόεδρο. Εδώ ακούσαμε τα διάφορα θέματα με τα οποία εσείς θέλετε να ασχοληθείτε. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία έκπληξη πολιτική για τις πόλεις, για την Ήπεθρο, διάφορα. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Αυτή η εδαφική συνοχή όσον αφορά το μέλλον, τι θα γίνει, ποιο ρόλο θα παίξει κανείς για μας το Κοινοβούλιο, πτυχή αυτή είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα συμβούν μετά από το 2013. Για τον κύριο Αντιπρόεδρο λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι οι προβλέψεις αυτά. Και το Μάρτιο, ναι, γνωρίζουμε ότι θα οργανωθεί η συνάντηση αυτή, νομίζω 26 Μαρτίου στη Δημοκρατία της Τσεχίας ίσως και ένα feedback στην Επιτροπή. Ε, αναφέρθηκε αυτή η πράσινη βίβλο. Θα πρέπει όμως να έχουμε μια λευκή βίβλο. Αυτό θα αποτελεί το πρώτο βήμα σίγουρα. Και έτσι θα έχει γίνει. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο, η κυρία Κρέλ έχει το λόγο. Äh, ναι, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να είμαστε τον πιο σύντομοι. Έχω κυρίως δύο ερωτήσεις. Πράγματι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε μια κρίση, πρέπει να είναι εξαιρετικές και οι αντιδράσεις μας όπως και τα γεγονότα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι το Συμβούλιο εδώ πέρα βρήκε έναν συμβιβασμό, το συζητήσαμε αυτό και στην ομάδα μας και θα το συζητήσουμε και στην Επιτροπή σήμερα το απόγευμα έτσι ώστε να παραμείνουμε στο πρόγραμμα, αλλά έχω εδώ πέρα ένα ερώτημα, όπως όλοι ξέρετε. Παραδείγματος χάρη, Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ το τι θα γίνει με την αλλαγή του κανονισμού του 2004 για την ενίσχυση της κοινωνικής στέγασης και μιλήσαμε για το τι θα γίνει για τα νέα κράτη-μέλη. Τώρα όμως έχει επεκταθεί αυτό και στα 27 κράτη-μέλη. Είναι μια κατάσταση που θα παγιωθεί ή είναι μια εξαίρεση, αν θέλετε, που εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Γιατί εδώ πέρα έχω μια παράξενη αίσθηση εγώ, γιατί δεν είχαμε και την δυνατότητα να το συζητήσουμε αναλυτικά αν είναι σωστό κάτι, τέτοια, ε, κάτι τέτοιο ή αν είναι κάτι το βραχυπρόθεσμο. Και εδώ πέρα συνδέεται άλλο ένα ερώτημα για αυτά με μένα. Μέχρι το... Υπάρχει αυτό το όριο του 4% των δαπανών που θα μπορεί να διατεθεί, αλλά είχαν προγραμματίσει αλλιώς τα κρατημέλη, είχαν υποβληθεί αλλιώς τα επιχειρησιακά σχέδια και δεν υπάρχουν νέα φρέσκα λεφτά, εάν κάτι σας κατάλαβα σωστά. Πώς θα το διαχειριστείτε λοιπόν αυτό. Δηλαδή το να εντάξει να κινηθεί γρήγορα Συμβούλιο Κοινοβούλιο Κομισιόν, αλλά τι θα γίνει όταν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα μετά από τα κράτη-μέλη στην πραγματικότητα. Πώς το βλέπετε, τι θα γίνει με τα επιχειρησιακά προγράμματα. Και ένα ερώτημα που ανέφερε ο κ. Τσούνεκ για την πρώτη προτεραιότητα, το μέλλον της πολιτικής συνοχής τι φαντάζεστε εσείς ότι θα γίνει, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή επιτάπητος και τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο όταν λέτε πως θα κάνετε τις πρώτες σας προτάσεις τον Απρίλιο σε μια σχετική διάσκεψη. Αυτό μπορεί να είναι καλό για την Προεδρία, αλλά είναι άσχημο για το Κοινοβούλιο, γιατί εμείς δεν θα είμαστε καν εκεί και αυτό με ενδιαφέρει για να δούμε τι μπορεί να κάνει ακόμα σε αυτή τη θητεία το Κοινοβούλιο. Αυτά σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μποπουή, συντονιστής από τους φιλελεύθερους. Κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε της Τσεχικής Προεδρίας, ε, εσείς μιλήσατε για το σχέδιο, για το φόρουμ, για τις ε, μακρινές περιφέρειές μας. Ε, νομίζω ότι θα εύκολο όμως να δειχθεί ότι θα πρέπει να πούμε τι πλούτο έχουν αυτές οι περιοχές για την Ευρώπη, γιατί συνήθως παρουσιάζονται σαν περιφέρειες που εντάξει χρειάζονται τα ευρωπαϊκά χρήματα, δεν δείχνουμε όμως τον πλούτο τους ή τουλάχιστον αρκετά ε, τα φυτά τους, τα ζώα τους, όλα αυτά που διαθέτουν και την γεωγραφική στρατηγική τους σημασία. Κρίμα που αυτά δεν τα παρουσιάζουμε, αλλά μόνο σαν περιφέρειες, σαν περιοχές που χρησιμοποιούν τα χρήματα τα ευρωπαϊκά, τα απορροφούν, δεν δείχνουμε όμως και τον πλούτο τους για τα ευρωπαϊκά κράτη, για την Ευρώπη ολόκληρη και ακόμα Κύριε Υπουργέ, το είχαμε συζητήσει την Παρασκευή που πέρασε στην Δημοκρατία της Τσεχίας στην Προεδρείο της Επιτροπής Περιφερειών, Παρασκευή πρωί για τον ε, εκστρατή αυτή που θα γίνει και θα δώσει τόσα πράγματα για το Μάρτιο που μας έρχεται. Θα πρέπει να δείξουμε ότι εδώ δεν πρόκειται για μια συζήτηση με μια αντιπαράθεση πέθρου και πόλης ανάμεσα σε τοπικές αρχές, περιφερειακές αρχές, κεντρικές αρχές. Θα πρέπει να δείξουμε πώς ε, σε μια συγκεκριμένη περιοχή τι μπορεί να κάνει ο πολίτης μεταφορές, τα κοινωνικά την απασχόληση, να κάνει κάτι σε αυτή την περιοχή, οποιαδήποτε είναι η πεθρος ή αστική περιοχή, γιατί συνδυάζονται, συνδέονται πολλές φορές αυτές οι περιοχές εντάξει. Όχι μία έκθεση που να δείχνει την αντίθεση ή να δείχνει νέες δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στις αρχές της εξουσίας εκεί, αλλά δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Το κύριο, το σιωφτικό εδώ, άμεσα τουλάχιστον όπως το είπαν και οι δύο συνάδελφοι, είναι αυτό το σχέδιο ανάκαμψης, αυτό το περίφημο σχέδιο ανάκαμψης για να τα συνδυάσω αυτά γιατί θα ασχοληθούμε και απόψε με την κινητικότητα σε αστικό επίπεδο, σε επίπεδο πόλεων. Θα δούμε στο ε, κοινωνικό ταμείο, στο περιφερειακό ταμείο να δούμε τι μπορεί να γίνει. Εδώ είχα απευθυνθεί τη Δευτέρα στο Στρασβούργο στην Επιτροπή που μας πέρασε και να πω ότι όσον αφορά αυτή την κινητικότητα υπάρχει μία αντίθεση στο πρόγραμμα δράσης. Θέλουμε κοινωνική ανάκαμψη και προγράμματα κοινωνικά, οικονομικά κλπ. Σε επόμενες εβδομάδες, ενώ από την άλλη μεριά να μην ξεχνάμε ότι ότι θυσιάζουμε πάρα πολλά ας πούμε, για θέματα ρήπανσης λοιπά Και θα δαπανίσουμε χρήματα για να βελτιώσουμε την κατάσταση για την ενέργεια και λοιπά στις κατοικίες, αλλά δεν κάνουμε τίποτα όσον αφορά την κινητικότητα σε επίπεδο πόλεων. Κρίμα. Κάτι ακόμα, θα έχουμε προκαταβολές, το είπατε αυτό και οι δύο σας. Είναι αυτές προκαταβολές, και το είπε ο κ. για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, εντάξει άλλαξε. Εμεί από το Κοινοβούλιο χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Εάν όμω απλά και μόνο διευκολύνουμε οικονομικά σκέτα τα κράτη-μέλη, όχι, διαφωνούμε. Και το τρίτο σημείο για αυτό το σχέδιο ανάκαμψης. Τώρα προχωράμε προς μια συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αυτό γίνεται και οι δύο συνάδελφοι προηγουμένως, κυρία Επίτροπε και κυρία Αντιπρόεδρο, σας είπαν ότι αυτό που ζητάμε στα κοινοβούλιο είναι να μπορέσουμε να σας συνοδεύσουμε και εμείς, αλλά υπάρχει ένας τέταρτος παράγοντας ε, εταίρος. Τα κράτη-μέλη, κύριε Επίτροπη, είπατε ότι ορισμένα κράτη-μέλη εντάξει είχαν κινητοποιηθεί, χαιρόμαστε γι' αυτό. Αυτό που θα θέλαμε σε ευρωπαϊκό κοινοβουλευτικό επίπεδο εδώ, εάν αυτό το Μάρτιο 27 υπουργοί από τις κυβερνήσεις να σας το επιβεβαιώσουν και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο παντού και στα τρέχοντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτοί θα κινητοποιηθούν. Εντάξει, δεν θα ήθελα τώρα να υπενθύμισω όλα πράγματα και θα ήθελα να σεβαστώ και το χρόνο, αλλά ορισμένα παραδείγματα σε διάφορες ε, χώρες δεν θα έχουμε αυτή την κατεπίγουσα εφαρμογή που απαιτείται και εγώ το λέω και το προτείνω στους συναδέλφους σχέση με τις ε, εκθέσεις που ψηφίσουμε. Εδώ τα κράτη-μέλη μεμονωμένα θα πρέπει να το επιτοπίσουν τι ευθύνε. Μην έλθουν εδώ τον Οκτώβριο που θα μα έρχεται ή το Δεκέμβριο εμεί φταίμε στι Βρυξέλλε και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, ό,τι όλοι φταίνε. Θα πρέπει ο καθένα σε αυτό το σχέδιο ανάκαμψη να αναλάβει τι ευθύνε του. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο από τη Φελευθερή Ομάδα και τώρα από του Πράσινου, ο κ. Κάλεμπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε για το ότι δεν μπόρεσα να ακούσω τις δηλώσεις ε, της κυρίας Επιτρόπου και του κυρίου Υπουργού. Είχε εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση το αεροπλάνο, αλλά τα ερωτήματα τα οποία θέσατε είναι... και αυτά τα οποία θα θέσω εγώ είναι παρόμοια με τον συναδελφον είπατε κύριε Επίτροπε flow as soon as possible. Και θα θυμάστε ότι πρόσφατα υπήρχε αυτή, αυτά τα παράπονα πως η διάθεση των κονδυλίων για την περίοδο 2007-2013 ήδη εν έτη 2008 ήταν πολύ περιορισμένα. Γι' αυτό έχω τις αμφιβολίες μου για το πώς θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Η κυρία Κρέλη ανέφερε πως ε, τα επιχειρησιακά προγράμματα επιβεβαιώθηκαν τον Ιούνιο 2008 και τώρα ξεκινάνε. Είπατε πως έχετε επισκεφθεί πέντε περιφέρειες, εάν όμως είμαι ε, σωστά πληροφορημένοι, έχουμε γύρω στις 260 περιφέρειες. Και δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ πέρα η σωστή προετοιμασία. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δηλαδή θα έχουμε πάλι άλλο ένα σχέδιο που θα βγάλετε από το σιρτάρι και θα είναι κατασκευή δρόμων. Τουλάχιστον αυτά ακούω από την ε, Γερμανία. Πράγματα τα οποία θα έχουν μόνο βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και δεν ξέρω εάν εκπληρώνουν και τις απαιτήσεις μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του κλίματος να συμφωνήσω εδώ πέρα βέβαια και με τον συνάδελφο για το σχέδιο αυτό δράσης για την αστική κινητικότητα και τελευταίο ερώτημα η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να ξανανοίξει τα επιχειρησιακά προγράμματα ίσως να κάνω λάθος αλλά θεωρητικά ίσως θα έπρεπε καθαρά θεωρητικά να ξαναδείτε και να επιβεβαιώσετε τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα. Και αν γίνει κάτι τέτοιο βράχει πρόθεσμα, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν γίνεται καν κάτι τέτοιο με το υπάρχον προσωπικό. Ευχαριστώ. Και για να ολοκληρώσουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων, θα ακούσουμε την κυρία Μποσίκοβα από τους Ανεξάρτητους. Κύρια Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αντιλαμβάνομαι ότι ήσταν πολύ ευέλικτοι όσον αφορά τις αντίδραση στην τελευταία οικονομική κρίση και αντιλαμβάνομαι και την ευελιξία των μέτρων που ελήφθησαν. Θα ήθελα εδώ πέρα λοιπόν να συμφωνήσω με τον κύριο Νίσελο και την κυρία Γκρέλ όσον αφορά το τι θα γίνει λίγο παρακάτω στο μέλλον. Τι άποψη έχετε για την πολιτική σε 2013, για να πάμε έτσι και σε ένα πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ευχαριστώ. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον Αντιπρόεδρο κ. Τσούνεκ. Λοιπόν, ε, συμφωνώ με την Επίτροπο για να δούμε ποιε... θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την Επίτροπο τι θα απαντήσει εκείνη, τι θα απαντήσω εγώ. Για να δούμε. Λοιπόν, θα απαντήσω σε όλες εκείνες τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το Συμβούλιο, που απευθύνεται και αφορούν το Συμβούλιο και ορισμένες ερωτήσεις, αυτές θα απαντήσει η Επίτροπος. Πρώτα απ' όλα, ο Βανίστελ Ρόι, ο κ. Βανίστελ Ρόι, ένα ερώτημά του. Τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος του προγράμματος αυτού, του νέου προγράμματος με τα έκτακτη στιγμή που απαιτεί έκτακτες ενέργειες, έχουν να κάνουν με τις θέσεις εργασίας, με το Ταμείο Λεγγύης και επίσης ε, κάτι που είχε ρωτήσει την κυρία Επίτροπο και εμένα με ρώτησε τι γίνεται με τη συνοχή, την εδαφική και την πράσινη βίβλο. Μερικές φορές μπορεί κανείς να απαντήσει ε, ταυτόχρονα και στις άλλες ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί και έτσι να επωφεληθώ όσο γίνεται περισσότερο από το χρόνο μιλίας που έχω στη διάθεσή μου. Λοιπόν, αυτό που έχει να κάνει με την πράσινη βίβλο που θα πρέπει αυτή να συμπληρωθεί, να καταλήξει, να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας αυτής. Να ολοκληρωθεί η συζήτηση, να περαθετωθεί η συζήτηση για την πράσινη βίβλο. Εντάξει θα μπορούσε να καταλήξει και σε μια λευκή βίβλο και έτσι θα μπορούσε να σας υποβληθεί. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν όροι για την νομοθεσία, για, συγγνώμη, για την διάρκεια αυτή της ε, θητείας του Κοινοβουλίου για το τι θα πρέπει να μπει στη Λευκή Βίβλο. Εσείς ξέρετε ότι απαιτείται μια κάποια περίοδος για την ολοκλήρωση της Πράσινης Βίβλου. Εδώ λοιπόν οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν στο μέλλον θα μπορέσουν να συνεχίσουν την παρακολούθηση αυτή. Θα αναφερθώ στην εδαφική συνοχή για το θέμα το οποίο το συζητάμε βασιζόμενοι σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε την κατεύθυνση την γεωγραφική που έχει σημασία και επίσης κάτι που μας αφορά από κοντά γιατί λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία τα οποία το καθορίζουν. Να σας πω κάτι, ποια είναι η πεποίθησή μου. Αυτό ακριβώς είναι και η συζήτηση στην Επιτροφή και για τους υπόλοιπους υπουργούς κλπ. Πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας αποκλειστικά αυτή την ε, γεωγραφική αρχή και τίποτα άλλο. Ταυτόχρονα χρειάζεται και μια εξέταση λεπτομερής ε, μεμονωμένα να δούμε τα διάφορα γεωγραφικά κριτήρια των περιφερειών και εδώ δεν αναφέρουμε μόνο για τις ε, περιοχές της μακρινές όπως αναφέρθηκε και ρωτήθηκε πριν από λίγο. Θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριληφθούν γιατί ακριβώς όλες και κάθε μία από αυτές τις περιοχές έστω και αν εξεταστούν αποκλειστικά γεωγραφικά για να δούμε αυτή τη διαφορά τους. Υπάρχουν, ε, επαναλαμβάνω, διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε μία περιοχή. Εντάξει, μια περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες από μια άλλη ορεινή περιοχή, στις Άλπεις ή ορεινή γενικά. Εδώ για αυτή την λευκή βίβλο, για την πράσινη βίβλο όπως αναφέρονται, υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλά ε, κίνητρα. Χρειάζεται να επωφεληθούμε από αυτή τη συζήτηση για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία που να συμπεριλαμβάνει και τη γεωγραφική αυτή αρχή ή τουλάχιστον να μην την αποκλεί και ταυτόχρονα να συμπεριλαμβάνονται και τα διάφορες αρχές, τα διάφορα κριτήρια για... που αναφέρονται από τους υπόλοιπους είτε είναι διάφορες πολιτικές και που να ισχύουν σε όλα αυτές τις περιοχές πολιτική σχετικά με την κρίση στις θέσεις απασχόλησης και διάφορα άλλα θέματα εκπαίδευσης, μόρφωσης κλπ. Αυτό είναι ένα θέμα ανοιχτό πάντως και γι' αυτό ακριβώς ε, τρέφουμε φιλοδοξίες. Επιθυμούμε η συζήτηση γύρω από την Πράσινο Βίβλο να ολοκληρωθεί, να περατωθεί υπό την δική μας τσεχική Προεδρία. Επίσης, ρωτήσατε κάτι. Εάν στο τέλος του προγράμματος αυτού, δεν ξέρω στην Επίτροπο, απευθήκατε σε μένα, Θέλετε να μάθετε αν θα ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα στο τέλος αυτού εδώ, είτε θα έχουμε μία αναθεώρηση του προγράμματος. Ποια είναι η απόψή μου και τα υπόλοιπα τα αφήνω για να τα απαντήσει η κυρία Επίτροπος. Εγώ θα ήθελα στην συμφωνία αυτή για νέα προγράμματα από το 2013, έτσι για να καταλαβαίνόμαστε, εδώ με μια συμφωνία για ένα νέο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν αυτή είναι δυνατή η συμφωνία, αν δεν εξετάσουμε πρώτα τι έχει γίνει, τι έχει συμβεί στην προηγούμενη περίοδο. Η Επιτροπή αναφέρθηκε σε διάφορες περιπτώσεις και εργάζεται υπό τον Γενικό Διευθυντή και όπως γνωρίζετε όταν ε, ειδωθήκαμε, συναντηθήκαμε στη Μασαλία, το συζητήσαμε. Εδώ έχουμε μια διευρυμένη επιτροπή για να εκπροσωπούνται όλα τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται να συλλογιστούμε γύρω από τα σημερινά προγράμματα. Τι σημαίνει η εργασία της Επιτροπής βέβαια να ολοκληρωθεί όσο γίνεται νωρίτερα το καλύτερο, το ιδανικό θα ήταν αυτό να γίνει υπό την Προεδρία τη δική μας και να όλα αυτά να τα εξετάσουμε πανσχάρι στα διοικητικό άχθος και σε διάφορα άλλα που έχουν να κάνουν με τα προγράμματα που ισχύουν και προωθούνται τώρα. Εγώ είμαι πεπισμένος, εάν η εργασία αυτή καταλήξει θετικά θα αποτελούσε μία βάση για τη νέα περίοδο προγραμματισμού τι εννοούμε ότι θα αλλάξει και ο σχετικός προσανατολισμός των πολιτικών όπως ακριβώς αναφερθήκατε εσείς για την εδαφική συνοχή από τη στιγμή βέβαια που θα ωφελήσει τα προγράμματα που θα υποβάλουμε και να λάβουμε υπόψη μας και την όλη διαχείριση τα καθεστώτα τα διάφορα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση που επικρατεί στις διάφορες περιφέρειες και με τον πρόεδρο. Δεν ξέρω, θα πρέπει να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις, σε όλους τους ευρωβουλευτές. Τι θα γίνει, θα, ή πώς θα πρέπει να απαντήσουμε έτσι γενικά. Εντάξει, κατ' επιλογή. Ωραία, μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τις απαντήσεις. Αλλά για να μην χάσω και το νήμα, να μην χάσω τη σειρά. Αναφερθήκατε ακριβώ για, το Ταμείο Αλληλεγγύης. Η κυρία Επίτροπος θα απαντήσει μάλλον. Να απαντήσω σε όσες ερωτήσεις αποτάθηκα σε μένα. Κύριε Λαμπερτ Βανίστερ Ρόι, αναφερθήκατε στην εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνάντηση με τους πολίτες. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες ε, για το τι θα αφήσει αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και προετοιμάζουμε και για την πολιτική συνοχή, ε, έγγραφα και πληροφορίες που να δείχνουν στους Ευρωπαίους πολίτες τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια για την πολιτική συνοχή για πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Επίσης έχουμε ετοιμάσει το για τις, για τις μεμονωμένες χώρες μέλη. Θα μοιραστούν στους Ευρωβουλευτές, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και στην επικοινωνία σας με τους πολίτες, με πολύ περισσότερες ε, πληροφορίες. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι και γι' αυτό συστήσαμε και την ε, ομάδα εργασίας για την απλούστευση. Και μαζί με την Προεδρία θα σας υποβάλουμε τα πορίσματα αυτής της ομάδας εργασίας που ελπίζουμε να μην σας απογοητεύσουν και να ενταχθούν και στο χρονοδιάγραμμά σας, να μην είναι εκπρόθεσμα. Ίσως στα τέλη Μαΐου μπορέσουμε να υποβάλουμε την έκθεση αυτή της ομάδα εργασίας, αλλά και νωρίτερα θα έχετε στοιχεία για την πορεία των εργασιών της. Ό,τι αφορά το Ταμείο ελληνικής προσπαθούμε με την ανακοίνωσή μας να κινητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη για να λάβουν υπόψη σοβαρά την ανάγκη αναθεώρηση του κανονισμού. Το αργότερο στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκριση αυτής της ανακοίνωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Κρέλ μίλησε για τις ε, κοινωνικές κατοικίες ε, σε σχέση με την ε, ενεργειακή απόδοση για τις εργατικές κατοικίες και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ανακοίνωση αυτή μιλά μόνο για ενεργειακή αποδοτικότητα και όχι για την ενεργειακή αποδοτικότητα σχέση με τη στέγαση με τις εργατικές κατοικίε. Μιλούμε περισσότερο για... Σίγουρα η στέγαση και οι κατοικίες είναι αυτέ που καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια, αλλά προσπαθούμε να βελτιώσουμε την απόδοση της ενέργειας και να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε και στην ε, ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού. Και αυτό το στόχο έχουν και οι τροπολογίες ε, δεν αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα εργατικών κατοικιών, αλλά μιλούν για τις κοινωνικές εισφορές που δίνονται στα κράτη-μέλη μέχρι 4% με στόχο να βελτιωθεί η απόδοση ενέργειας και να χρησιμοποιηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη στέγαση. Θα εξαρτηθεί όμως από τα κράτη-μέλη να επιλέξουν τι είδους ε, ε, στέγη θα χρησιμοποιήσουν για την ε, νέα αυτή δυνατότητα. Δεν υπάρχουν ε, νέα κονδύλια, χρησιμοποιούμε τις ε, ισχύουσες εισφορές. Απλώς προβαίνουμε σε μία μετατόπιση, σε μία αλλαγή του συνήθους τρόπου δαπανών και του καταμερίσμου, γιατί συνήθως η απορρόφηση είναι πολύ αργή δεν ξεκινά από την πρώτη μέρα του προγράμματος, γιατί χρειάζεται μια προεργασία, μια ολοκλήρωση του προγράμματος, μια διαδικασία ελέγχου, προκειμένου το σύστημα αυτό να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Αυτό που προσφέρουμε λοιπόν στα κράτη-μέλη είναι μια δυνατότητα να μετατοπίσουν ένα τμήμα των κονδυλίων που κανονικά θα χρησιμοποιούνταν σταδιακά κατά το δεύτερο ημισή του περίοδου, να το μεταθέσουν στις ε, συμπληρωματικές ε, προκαταβολές ε, για τις φετινές δαπάνες, επιταχύνοντας τις δαπάνες αυτές μέσω και της συρρήκνωσης του διοικητικού άχθους και χάρη και στην εφαρμογή των τροπολογιών του κανονισμού για να διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πρόσβασή τους στα κονδύλια προκειμένου οι, τα κονδύλια της τις να εκταμιεύονται με ταχύτερους ρυθμούς. Δύο φορές τέθηκε το ερώτημα πάλι για την απόδοση αυτού του προγράμματος και το ρυθμό εκταμίευσης. Να συνεχίσω εγώ, λέει ο Τσέχος Αντιπρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη γιατί ήμουν λίγο ασυνάρτητος προηγουμένως στις απαντήσεις μου, ανοργάνωτος. έπρεπε να είμαι πιο συγκροτημένος. Ξέχασα την ερώτηση για τη στέγαση, γιατί η ερώτηση αυτή είχε υποβληθεί πριν τη μετάβαση από το 2% στο 4%. Ε, είναι 2 συν 4, δηλαδή η παρούσα κατάσταση έχει ως εξής. Στα προγράμματα έχουμε ένα 2% που μπορεί να παραχωρηθεί για τη στέγη, αλλά αυτό το 2% δεν έχει σχέση με το 4% που ανέφερα εγώ στην ε, ομιλία μου, που είναι μια συμπληρωματική ε, πρόταση. Αυτό το 4% αναφέρεται στις επιδοτήσεις, ε, στα κονδύλια που έχουν τα κράτη-μέλη για την περίοδο 2007-2013. Και αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή δεν είναι συμφωνία. Όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κονδύλια αυτά. Προηγουμένως η εκπρόσωπος των Πρασίνων με ρώτησε αν ε, θα ισχύσει αυτό για πάντα. Τα μέτρα αυτά είναι έκτακτα γιατί αντιμετωπίζουμε και μια ενεργειακή κρίση. Για την θέρμαση των κατοικιών, τα κράτη-μέλη χρειάστηκε να αυξήσουν το ποσοστό Είναι το 15% περίπου η στέγη των κατη... των κατοικιών τη συνολική κατανάλωση τη ενέργεια ενό κράτου. Πάνω κάτω, ανάλογα και με τι διαστάσει του κράτου. Στόχο μα όμω είναι να έχουμε μια εξοικονόμηση τη ενέργεια και είμαστε ελπισμένοι ότι με την υιοθέτηση αυτή τη απόφασης ε, θα σημειώσουμε πραγματική πρόοδο και θα ωφελήσουμε όλους τους δικαιούχους χωρίς να δημιουργήσουμε νέους ε, θερμοελεκτρικούς σταθμούς ή νέα εργοστάσια και ταυτόχρονα μειώνοντας τις δαπάνες, ενεργειακές δαπάνες των Ευρωπαίων πολιτών. Με τα μέτρα αυτά, με αυτό το συμπληρωματικό 4% θα μπορέσουν τα κράτη-μέλη, το καθένα ξεχωριστά, να βρουν τα καλύτερα προγράμματα, να διαλέξουν μέσα από ένα φάσμα προγραμμάτων για την περίοδο αυτή και έτσι να αποφασίσουν ποια είναι τα καλύτερα προγράμματα και να επιλέξουν αυτά που τους ε, ικανοποιούν και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Αυτά θα ήθελα να πω συμπληρώνοντα την ε, απάντηση της Επιτρόπου. Αυτά για το πακέτο που στόχο έχει τη βελτίωση των κατοικιών. Παραμένει λοιπόν το 2% για τα νέα κράτη-μέλη. Είναι άσχετο με το 4% που θα ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτά ε, λοιπόν για το θέμα της ε, στέγασης. Πολύ καλά. Έχουν ζητήσει... πέντε συνάδελφοι τον λόγο. Παρακαλώ σύντομα σύντομα για να προλάβουν όλοι να λάβουν τον λόγο. Συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρεζίνα. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου απαντήθηκε ήδη εν μέρη από την κυρία Επίτροπο και τον κύριο Υπουργό γιατί ήθελα να σας ρωτήσω τι θα κάνατε για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ε, στέγασης. Οπότε σας ευχαριστώ για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στήλερ. Κυρία Στήλερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως. Κυρία Επίτροπε, ε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει κρίση, άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους και πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξαναβρουν δουλειά. Αυτό είναι το νόημα των διαρθρωτικών ταμείων. Μιλήσατε για την ηλιακή ασφάλεια και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν ε, δουλειές. Θέλω να μου πείτε εσείς ποια θεωρείτε ότι ε, είναι η δυναμικότητα της πράσινης οικονομίας και των πράσινων θέσεων εργασίας αυτό το οποίο ακούστηκε το όνειρο του Ομπάμα στην Αμερική οπότε ήθελα να ακούσω κάποια πράγματα περισσότερα αναφέρατε την κοινωνική στέγαση και το ότι δεν υπάρχει ορισμός είναι έσχος το ότι δεν έχουμε ακόμα ορισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή φτώχεια και την φτώχεια καυσίμων κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα επίσης για την απλοποίηση και την ε, απόδοση ευθυνών και τη λογοδοσία. Πράγματι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε προς σωστή κατεύθυνση, να υπάρχει μια σωστή ε, σωστός υπολογισμό και να ξέρουμε που πηγαίνουν τα χρήματα προλογουμένου. Θεωρείται πως πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πιο τυπική και γραπτή ως προς αυτό. Ευχαριστώ και τους δύο λοιπόν που ήλθαν εδώ και μας ε, λένε όλα αυτά και σε όλους ε, τους συναδέλφους μας λένε για το μέλλον της Επιτροπής της ε, πολιτικής συνοχής ε, και για το πρόγραμμα ανάκαμψης, για την περιφερειακή πολιτική. Όλα αυτά τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης. Δεν θα υποβάλω κανένα ερώτημα επειδή δεν έχουμε χρόνο και επειδή έτσι και στη συνέχεια θα διεξαχθεί μια συζήτηση. Απλά και μόνο υποβάλλω ερώτημα το οποίο σας έχει υποβληθεί και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει περισσότερο εργό ρόλο προ την κατεύθυνση αυτή. Γνωρίζουμε ακριβώ ότι μπροστά αυτή την κατάσταση, αυτή τη σημερινή, εδώ χρειάζεται να είναι κάνει γοργός. Ε, είναι απαραίτητο αυτό και θεωρούμε ότι σε αυτή τη διαδικασία για να πετύχουμε μια τελική συμφωνία το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να παίξει ένα περισσότερο εργό ρόλο και έτσι καλλιώς ε, θα πρέπει να τον παίξει αυτή τη στιγμή για να ελπίσουμε και να πετήσουμε και στο μέλλον επίση, εδώ στην ομάδα εργασία να να αυτά σε σχέση με αυτές τις ε, διαδικασίες απλοποίησης των κανονισμών. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα μπορούσαν να παίξουν ένα περισσότερο σημαντικό ρόλο, πρωταγωνιστικό από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Τουλάχιστον έτσι αλλιώς γνωρίζουμε ε, την ανάγκη να προωθηθούν αυτές τι πρωτοβουλίες και αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που περνάμε τώρα το Κοινοβούλιο ε, ε, δεν θα πρέπει να είναι κάτι που θα αναχαιτίζει την όλη πορεία για να αποφύγουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Αντίθετα θα πρέπει να παίξει θετικό ρόλο για την πολιτική συνοχή και για την πράσινη βίβλο. Η περιφερειακή ανάπτυξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και υπάρχει μια έκθεση που ολοκληρώθηκε από τον κύριο Βανίστερ Ροέ και που είχε ιδιαίτερη απήχηση. Είχαμε και πάνω από 200 τροπολογίε από του συντρόφου ε, και τη επιτροπή από τους συναδέλφους ε, και νομίζω ότι ε, έχει σημασία πραγματικά η πράσινη βίβλος και να ζητήσουμε και από τους δύο να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που έχουν γεννηθεί πάνω σε αυτό. Αυτές τις στιγμές έχει ξεκινήσει μια περίοδος διαβουλεύσεων και θεωρώ ότι σημαντικό θα ήταν από τη στιγμή που θα περατωθεί αυτή η διαδικασία και θα ακούσουμε τους διάφορους εταίρους και όσοι συνεργάζονται για την, Επιτροπή, για την Πολιτική Συνοχή και για το ρόλο του Κοινοβουλίου, τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες, την κοινότητα πολιτών. Από τη στιγμή που θα έχουμε έχουμε ακούσει όλους αυτούς ε, να μπορέσουμε να μεταβιβάσουμε αυτήν την ιδέα. Τι αντίληψη έχουμε σχετικά με αυτήν τη συνοχή, την εδαφική και ε, ε, αρκετοί μας λένε ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Σημαντικό είναι να το έχουμε καταλάβει ότι αυτή η πολιτική εξελίσσεται. Βλέπουμε πώς προχωρούν οι διάφορες περιφέρειες προς μια συνοχή. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα σε μια διαπεριφερειακή, ενδοπεριφερειακή συνοχή και τις διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες. Τις βλέπουμε, τις βλέπουμε καθαρά και θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα οικονομικά μέσα που διαθέτουμε τώρα και έτσι αυτές οι διαφορές μέσα σε αυτές τις περιφέρειες να γίνουν όσο ένα και λιγότερο μικρότερες. Ο κ. Σαραγκόσο, στη συνέχεια δε ο κ. Αγγελάκας και ολοκληρώνουμε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και τη Συμβούλιο και την Κομισιόν για το έργο τους και την συνεισφορά τους με τις γρήγορες αυτές ε, λύσεις που προτείνουν αυτή τη στιγμή. Θεωρώ πως οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν όμως κάποια ερωτήματα που έχουν τεθεί και θα ήθελα να τα θίξω. Είπατε πως πρώτος και κύριος στόχος είναι να δοθεί μια τονοτική ένωση στην ε, ευρωπαϊκή οικονομία και ένας τρόπος ε, είναι να χρησιμοποιηθούν και τα ταμεία συνοχής για την ε, στέγαση και να χρηματοδοτηθεί η οικονομική αποδοτικότητα. Βέβαιω, εάν να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη για αυτό το στόχο, για την στέγαση πρέπει να υπάρχει κάποια ως ένα προσανατολισμός και δεν ξέρω εάν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε εγκαίρω και γρήγορα όπω λέμε και δεν ξέρω αν θα έπρεπε εδώ πέρα να προσθεθούν και οι φτωχότερες περιφέρειες Ευρώπης σε αυτή την χρηματοδότηση για να εκλείψουν οι παραγκουπόλεις και τα γκέτο το οποίο χρειάζεται και η χώρα μου, η Ουγγαρία ιδιαίτερα. Δεύτερον ερώτημα, πώς θα εφαρμοστεί συγκεκριμένα αυτή η πρόταση, πώς θα προτεθεί στις υπάρχουσες προτάσεις. Και τρίτον, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά κανόνα χρηματοδοτούνται μόνο μέτρα ενεργούς απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή όμως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τις ε, δουλειές τους, οπότε θα έπρεπε για μια μεταβατική περίοδο να χρησιμοποιηθούν και παθητικά μέτρα. Τέλος, ε, καταλήγεται με μια πρόταση που μιλάει για δαπάνες που δεν είναι ε, μισολογικές και ότι θα πρέπει να κοπούν γιατί αυτό έμεινε έξω από τις ε, προτάσεις του Συμβουλίου και είναι δυνατόν να ξαναπροσθεθεί ο κύριος Αγγελάκας. Ευχαριστώ και τον κύριο Κούνεκ και την Επίτροπο για την ενημέρωση που μας έκαναν. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Τσεχική Προεδρία. Ε, είμαι εισηγητή στην ε, τροποποίηση του κανονισμού 1080. Επί της ουσίας θα μιλήσουμε μετά στην κουβέντα που θα κάνουμε. θεωρώ σωστή την κίνηση της Επιτροπής του Συμβουλίου να τροποποιήσουν αυτούς τους τρεις κανονισμούς ε, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες ανάγκες, την έκτακτη κρίση που υπάρχει. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, ψάχνοντας τα στοιχεία για να δω κατά πόσον ο κανονισμός 1080 του 2006 αξιοποιήθηκε από την ημέρα που ψηφίστηκε μέχρι σήμερα, είδα ότι το ποσοστό απορρόφησης από τα νέα κράτη-μέλη, όπως λέγονται, ήταν πάρα πολύ χαμηλό, κάτω από 1%. Λέω λοιπόν εν μια υπόθεση ότι σε δύο μήνες έχουμε τροποποιήσει τους κανονισμούς. Θα ήθελα να ξέρω ποιο πρόγραμμα παρακολούθησης της υλοποίησης έχετε σκεφτεί, πώς ε, θα, πιέσετε τα κράτη-μέλη να βγουν γρήγορα και να υλοποιήσουν αυτές τις ε, τροποποιημένες διατάξεις, ούτως ώστε να μην χαθεί χρόνος πολύτιμος, τα χρήματα να πάνε σε αυτούς που πρέπει να πάνε και κατά πόσον σκέπτεστε να ενημερώσετε και την Επιτροπή μας πάνω στην πορεία υλοποίησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα στα ερωτήματα τα οποία ίσως ε, παραλείψαμε στον προηγούμενο γύρο. Νομίζω πως ξέχασα να απαντήσω στην ερώτηση για τη σχέση μεταξύ πόλεων και υπαίθρου. Κατά την άποψή μας σε πολλά ε, κράτη-μέλη ο λόγος, η σχέση ανάμεσα στις πόλεις και την Ήπεθρο είναι 95 προς 5, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις 75 με 25. Ε, σαφώς λοιπόν είναι προς το συμφέρον μας ε, να διασφαλίσουμε πως οι πολίτες ε, θα μπορούν να συνεχίσουν να ζουν εκεί που ζουν αυτή τη στιγμή υπό την προπόθεση πως η ποιότητα της ζωής τους και της στέγης τους ε, θα διατηρείται για να έχουν και κίνητρο να μείνουν εκεί που μένουν και όχι να αναγκάζονται να φύγουν. Το θέμα δεν είναι μόνο χρηματικό, είναι και θέμα επιλογής ενός τρόπου ζωής. Αν κάποιος ζει σε μια πόλη και χρειάζεται 20 λεπτά να πάει με τα πόδια σε ένα νοσοκομείο, για να έχει τις ίδιες συνθήκες ε, με κάποιον ο οποίος ζει 100 χιλιόμετρα μακριά από μια πόλη ε, όσον αφορά λοιπόν τις ε, βασικές ανάγκες πρέπει αυτές να καλύπτονται ανεξαρτήτως με του που μένει ο καθένας θέλουμε λοιπόν οι σχέσεις ανάμεσα της πόλης και την υπεθρό να είναι ισορροπημένες, τουλάχιστον στο βαθμό που να μπορέσουμε να εμποδίσουμε αυτή την έξοδο των ανθρώπων από την Ήπεθρο προς τις πόλεις. Και σε κάποιες χώρες το έχουμε επιτύχει. Σε άλλες χώρες ε, υπάρχουν ε, τα προάστια αυτά γύρω-γύρω από τις πόλεις ε, και ο κόσμος φεύγει από τα κέντρα των πόλεων, φεύγει από τις πόλεις, μένει κοντά στις πόλεις μεν, αλλά ε, στην ύπεθρο Δεν θέλουμε ε, αυτό το πράγμα. Εμείς, εμείς θέλουμε όπου και να μένουν οι άνθρωποι να έχουν ε, μια συγκεκριμένη ποιότητα ζωής. Και βεβαίως τι θα κάνουμε τώρα για να μπορέσουμε να παραγκάσουμε θέλετε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτά τα ε, προγράμματα και τι θα γίνει και με το 4% αυτό το οποίο δίνουμε τα κονδύλια εάν η απορρόφηση δεν είναι αρκετά υψηλή. Το να μπορέσουμε να εγκαλέσουμε ένα κράτος μέλος ε, είναι κάτι το πολύ δύσκολο σε περίπτωση παραδείγματος χάρη που δεν προωθεί την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Εμείς θεωρούμε απλά πως είναι τόσο γενναιόδορη η προσφορά μας που πραγματικά δεν θα την προσπεράσουν τα κράτη-μέλη, θα την ε, χρησιμοποιήσουν. Και βεβαίως ε, το ποσοστό αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε από έναν διάλογο και για να απαντήσω εδώ και στην συνάδελφο των ε, Πρασίνων πρόκειται για ένα μόνο από τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας και που θα έχουμε μετά το 2013. Με βάση την ε, εμπειρία μας ίσως ε, να ευνοηθεί πράγματι η εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε βεβαίω για την μόνωση κτηρίων, αλλά ταυτόχρονα χρηματοδοτούμε και ηλιακού συλλέκτες και τέτοια πράγματα. Όλα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν με το 4%. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα πως η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει με τα έργα αυτά εξοικονόμησης ενέργειας και να κινητοποιηθεί περισσότερο σε αυτό το τομέα. Άκουσα εδώ πέρα κάποια κριτική πως η Ευρώπη δεν μπορεί να ορίσει την κοινωνική στέγαση. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί ευρωβουλευτές που δεν ασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα στην καριέρα τους και αν όλοι μαζί καθίσουμε και δούμε ο καθένας τον ορισμό που έχει για την κοινωνική στέγαση δεν νομίζω ότι θα είναι ταυτόσιμη. Και βεβαίω γιατί σημαίνει αυτό. Γιατί διαφορετικές περιφέρειες έχουν διαφορετικό επίπεδο προστασίας και γι' αυτό ακριβώς είμαστε μια Ευρώπη των περιφερειών. Υπάρχει και διαφορετικό επίπεδο, διαφορετικός μέσος όρος εισοδήματος, διαφορετικό ποσοστό του εισοδήματος ξοδεύεται στην ε, στέγαση, στις ε, διάφορες περιφέρειες. Όλα αυτά επηρεάζουν τον ορισμό της ε, κοινωνικής στέγης. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε Νομίζω λοιπόν πως ε, έχουμε λίγο υστερήσει προσπάθειές μας ε, ως προς αυτό. Πρέπει να βρούμε μια εφικτή απόφαση και θεωρώ πως ε, δεδομένου του ότι έχουμε και 27 χώρες και πολύ περισσότερες περιφέρειες κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη και όταν φτάσουμε σε παρόμοιο επίπεδο των περιφερειών θα είναι και ευκολότερο να συμφωνήσουμε στον ε, ορισμό αυτόν. Θα να ευχαριστήσω την κυρία Περέζ για το ερώτημά της για την ε, Λευκή Βίβλο. Η Επίτροπος βεβαίω ε, ήταν αυτή που έκανε το μεγαλύτερο έργο σε αυτό τον τομέα και θα ήθελα να την ευχαριστήσω. Και μάλιστα ε, ήταν κάτι το οποίο απαιτούσε θάρρος να προσπαθήσει δηλαδή να ορίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν και να μπουν σε μια λευκή βίβλο και νομίζω πως ε, τα αποτελέσματα θα τα δούμε σε δύο-τρεις μήνες από τώρα όταν θα συζητήσουμε την ε, Λευκή Βίβλο και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Επίσης θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Βοποσίκοβα για την ανάπτυξη αυτής της πολιτικής μετά το 2013. Εγώ είμαι πεπισμένος πως θα αναπτυχθεί διαφορετικά από ό,τι σκεφτόμασταν πριν από έξι μήνες. Είναι τόσο μεγάλης η προκλήση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η ενεργειακή ε, ανεξαρτησία που είναι τόσο πλέον οξυμένη ως ανάγκη που δεν γίνεται παρά να επηρεάσει την πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Όλα αυτά βεβαίως ε, συνδέονται και με τις ε, νέες προκλήσεις που έχουμε το νέο έτος και όποτε μιλάμε, με συναδέλφους βλέπω πώς αλλάζουν οι νοοτροπίες και βεβαίως παρά το ότι εξακολουθούμε να θέλουμε να δώσουμε ένα πιο ισόρροπο επίπεδο, ένα πιο ισόρροπο επίπεδο ανάπτυξης στην, ε, στις περιφερειές μας ε, ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη και η ε, αλληλεξάρτηση εντό Ευρώπη και η εξοικονόμηση ενέργεια. Τώρα για το ερώτημα του Ούγγρου βουλευτή, ίσως να μην σα αρέσει η απάντησή μου. Με ρωτήσατε για το εάν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να χρησιμοποιηθεί και για έμεσες πληρωμές. Κοιτάξτε, βασικά όταν τέθη αυτό το ζήτημα υπήρχε μια θεμελιώδης διαφωνία. Νομίζω πως η Ουγγαρία ήταν απομονωμένη. Και πραγματικά δεν θέλω τώρα να σας δώσω εδώ πέρα ελπίδες ε, που δεν έχουν βάση ότι θα αλλάξουν δηλαδή τα πράγματα στο μέλλον. Και ο λόγος είναι απλός. Τα λεφτά είναι μετρημένα. Και άρα το 4% ακόμα και η προκαταβολή το 2,5% για όλα τα κράτη-μέλη, συν το 2% το επιπλέον για τα νέα κράτη-μέλη, όλα αυτά είναι εις βάρος της κατανομής που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο προϋπολογισμός, ο διαθέσιμος δεν αλλάζει. Οπότε, αυτά ε, ως απάντηση. Ε, σε αυτά θα μείνω, δεν ξέρω αν δεν απάντησα κάτι. Να διευκρινίσω κάτι που Ρωτήσατε και προηγουμένω για το βαθμό απορρόφηση σε αυτή τη φάση των δημοσιονομικών προοπτικών. Εμείς ε, προσδιορίζουμε την απορρόφηση με ένα σχετικά πρωτόλιο μέσο που είναι η διάμεση πληρωμή που στηρίζεται στην ε, επιστροφή ουσιαστικά. Είναι λογικό που σε αυτή τη φάση η εκταμείευση από τις ενδιάμεσες πληρωμές ε, θα δοθούν μετά την υιοθέτηση τη αξιολόγηση ε, συμμόρφωση. Γι' αυτό και είναι χαμηλό το ποσοστό απορρόφηση αυτή τη στιγμή. Και αυτό ισχύει γιατί είναι μια πολιτική που στηρίζει στι επιστροφέ και έχει και προκαταβολές. Αν εγκριθούν οι τροπολογίε αυτές στον κανονισμό, οι προκαταβολές για τις τρεις χρονιές 2007, 2008 και 2009 για τις 15 χώρες θα φτάσει 7,5% των ε, κονδυλίων χώρες και 9,5% για τις νέες χώρες. Περίπου στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ όλα μαζί. Οπότε η δική μας πρόκληση, όπως ε, είπε και ο Ζαν Μαρή Παπουή, είναι να εξασφαλίσουμε να μην μένουν οι προκαταβολές στα ταμεία, αλλά να φτάνουν στους δικαιούχους, προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις και να ε, συμβάλλουν αυτές οι προκαταβολές σε μια όθηση των ε, επενδύσεων, σε μια προβολή των επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την νομική ίσια για να επιβάλλουμε αυτά τα μέτρα στα κράτη-μέλη, αλλά συνεχίζουμε τις εργασίες και επισημαίνουμε την ανάγκη της χρησιμοποίησης των προκαταβολών με τρόπο που να συμβάλλει στην αύξηση των επενδύσεων, στην τόνωση των επενδύσεων και να φτάνει γρήγορα στους δικαιούχους. Επίσης, συμφωνώ με την κυρία Γκαρθία Πέρες ε, επειδή σπεύσαμε να ανταποκριθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στην κρίση, πέρασε με εξαιρετική ταχύτητα αυτός ο κανονισμός, κάπως βεβαιασμένα, και συμφωνώ ότι για τις περαιτέρω απλουστεύσεις θα είναι χρήσιμη και η συνεργασία και θα φέρει και καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί σπουδή μερικές φορές είναι κακό σύμβουλος. Το έργο του Συμβουλίου και τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου ε, οδήγησαν σε μία άτυπη έγκριση του κανονισμού σε επίπεδο κορεπέρ πριν τα Χριστούγεννα. Ήδη το Συμβούλιο έχει εγκρίνει τις αλλαγές στο Γενικό Κανονισμό, κάτι που μας ε, επιτρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, της ε, σύμφωνης ε, γνώμης για να εμπλέξουμε και το Κοινοβούλιο. Και χαίρομαι που το Συμβούλιο έδρασε τόσο ε, ακαριέα και θα μπορέσουμε να έχουμε την έγκριση του κανονισμού εμπρόθεσμα. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο δυναμικό της πράσινης οικονομίας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στις κλιματικές αλλαγές την ανάγκη μετριασμού τους, αλλά δεν ε, δίνουμε αρκετή έμφαση στο δυναμικό δημιουργής θέσεων απασχόλησης που ενέχει, εμπεριέχει αυτή η πράσινη οικονομία. Πριν από τρία χρόνια δώσαμε 9 δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, απόδοση της ενέργειας και την ε, προαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και ήδη δρεύουμε τους πρώτους καρπούς της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Τον Ιούνιο θα έχουμε την βαλαιοσκαδιναβική συνδιάσκεψη για τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργεί η ενεργειακή απόδοση και ο οικολογικός χαρακτήρας της οικονομίας. Νομίζω έτσι θα μπορέσουμε να σκεφτούμε και υπό διαφορετικό πρίσμα και τις κλιματικές αλλαγές. Επίσης, προσοχή, απλούστευση δεν σημαίνει καταστρατήγηση των δημοσιονομικών ε, κανόνων ή χαλάρωση των ελέγχων. Επουδενή δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Δεν σημαίνει ξέφραγο μπέλη ε, απλούστευση. Απλώς ε, με την απλούστευση μειώνεται η πιθανότητα λάθους, γιατί πολύ συχνά οι περίπλοκες και πολυσύντες διαδικασίες οδηγούν σε σφάλματα εξαιτίας του δυσεφάρμοστου χαρακτήρα τους. Έτσι με την απλούστευση θα μειωθούν τα λάθη αλλά αυτό θα γίνει με σεβασμό των δημοσιονομικών κανόνων. Η προσέγγιση μας δεν πρόκειται να προσβάλλει, να καταστρατηγεί τους κανόνες αυτούς. Επίσης έχω και ένα γενικό σχόλιο. Μιλούμε τώρα για κανονισμό Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, ε, αλλά υπάρχει και κανονισμός της Επιτροπής, που θα αναθεωρηθεί αμέσως μετά την έγκριση της αναθεώρησης του κανονισμού του Συμβουλίου. Και χάρη στι τροπολογίε αυτές, ε, χάρη στι αλλαγές που θα γίνουν στο κανονισμό του Συμβουλίου, θα επηρεαστεί και ο κανονισμός ε, τη Επιτροπή και θα δούμε πώς θα βελτιωθεί και εκεί η απλούστευση και η διευκόλυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό ταμείο, αν κατάλαβα καλά, τα κράτη-μέλη αλλά και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Επιτροπής θεωρούν ότι θα γίνει μια σημαντική μεταστροφή στη φιλοσοφία του κοινωνικού ταμείου αν υιοθετηθεί αυτό το μέτρο, αλλά θα πρέπει να το εξετάσουμε πιο διεξοδικά. Αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό σίγουρα. Σήμερα μίλησα περισσότερο για επιτάχυση των διαδικασιών παρά για μεταστροφή στη φιλοσοφία μας. Σε ό,τι αφορά τον αναπρογραμματισμό, αν γίνει ε, αναπρογραμματισμός παντού είναι κάπως δύσκολο, γιατί θα ανοίξουν σίγουρα κάποια προγράμματα, γιατί ορισμένες χώρες δεν έδωσαν έμφαση σε συγκεκριμένα θέματα που πια είναι κρίσιμα και φλέγοντα δεδομένες κρίσης που διανύουμε. Πάντως θέλουμε να μεριμνήσουμε ώστε να μην ε, αλλάξουμε την πορεία μας που θα μας φέρει σε μια πιο πράσινη οικονομία, σε μια πιο ανταγωνιστική και καινοτόμα ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν θέλουμε να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με τους στόχους αυτούς, απλώς θέλουμε στα προγράμματα να βελτιώσουμε τον αντίκτυπό τους στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη χρήση των υποδομών, στην ενέργεια και εκεί θα έχουμε επαφές με κράτη και περιφέρειες και με τους αρμόδιους για τα θέματα αυτά και θα συνεργαστούμε. Σας είπα ότι τελευταία, το τελευταίο δεκαήμερο επισκέφθηκα πέντε περιφέρειες. Αυτό φέτος όμως. Αλλά γενικώ ε, έχω επισκεφθεί 240 από τις 271 περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα δεν ήταν να πω απλώς ότι πέντε περιφέρειες συμφωνούν, γιατί συνεργαζόμαστε με όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και όλοι οι αρμόδιες περιφέρειες γνωρίζουν το δυναμικό αυτό. Γι' αυτό και περιμένουν να εγκριθεί για να το εφαρμόσουν. Πάντως, όπως είπε και ο Υπουργό, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε εμείς είναι να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Γι' αυτό και εσείς θα μπορούσατε να συμβάλλετε προκειμένου να εφαρμοστεί και στην πράξη αυτό το τεράστιο δυναμικό που δημιουργείται και να αξιοποιηθεί. Θα γίνει ένα προγραμματισμός, το συντομότερο δυνατό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν στρατηγικό χαρακτήρα, δεν είναι λεπτομεριακά προγράμματα. Δεν χρειάζεται αναπρογραμματισμός να γίνει παντού. Δύο τρίτα των επιχειρησιακών προγραμμάτων χρειάστηκαν παράταση για την αξιοποίηση του δυναμικού. Και το πρώτο εξάμεινο του έτος θα έχουμε τις επενδύσεις από την αξιοποίηση των υφισταμένων προγραμμάτων. Αυτά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ξεπεράσαμε το χρόνο που είχε προβλεφθεί, αλλάξιζε τον κόπο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο προσκεκλημένους μας και να ολοκληρώσουμε με το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης ε, συνοψίζοντας ως εξής. Τώρα ακριβώ θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων για τις εκθέσεις ε, για τη, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής και εδώ σχετικά με τον κανονισμό του Κοινωνικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για τάξη περί δημοσιονομικής διαχείρισης. Και αν συμφωνείτε και οι συντονιστέ σήμερα το απόγευμα και στη συνέχεια το σύνολο της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής να προβλέψουμε η Επιτροπή μας να μπορέσει να ψηφίσει και αυτό σε μια έκτακτη συνάντηση για τις 9 Μαρτίου και έτσι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσει ε, και του χρονιογράμματος από πλευράς Επιτροπής και Συμβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο σας για την παρουσία σας ανάμεσά μας. αγαπητοί συνάδελφοι, έχει προχωρήσει η ώρα και πρέπει να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας, οπότε περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής Διατάξης περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης, η η κυρία Γκαρσία Πέρες, οπότε της δίνω τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο προηγούμενο σημείο κάνα μια συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις αυτές για αυτές τις αλλαγές για τις διατάξεις των κανισμών και κάτω από τη σημερινή οικονομική κρίση. Και τότε γνωστοποίησα την άποψή μου Παρακαλούμε λίγη ησυχία. Λοιπόν, τη ε, διάθεση αυτής της Επιτροπής ε, να συμμετάσχει περισσότερο ενεργά στην προ... υποβολή αυτών των προτάσεων. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο ιδιαίτερα, αλλά εδώ να ενημερώσουμε τους συναδέλφους ότι είναι σύμφωνη γνώμη εδώ στα πλαίσια αυτά βρισκόμαστε δεν έχουμε δυνατότητα έστω και αν είχαμε τη διάθεση έστω και αν όλοι μας συμφωνούσαμε να επιφέρουμε κάποια αλλαγή σε αυτή τον κανονισμό δεν την έχουμε. Τη μόνη δυνατότητα που διαθέτουμε είναι να πούμε ή όχι αν συμφωνούμε και όπως μας είπε και η Επίτροπος, μας εξέπληξε η ταχύτητα με την οποία πέτυχαν πάνω σε αυτό όλα τα κράτη-μέλη μια συμφωνία. Αυτός ο οργανισμός τι κάνει, επιταχύνει αυτή τη διαδικασία ώστε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στη διαχείριση και του Ταμείου Συνοχής και της Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω περισσότερων προκαταβολών με διάφορες άλλες δυνατότητες, ε, διάφορες προσπάθειες διαχείρισης ε, κατάλληλης των ταμείων ε, και για τα γενικά έξοδα να είναι υποχρεωτικά όπως είπαμε και διάφορα θέματα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, θέματα που έχουν να κάνουν με τις προκαταβολές των πληρωμών όλα αυτά. Εδώ Εάν τα συζητούσαμε βέβαια πάνω στορισμένα θα συμφωνούσαμε περισσότερο από ό,τι με άλλα. Από ό,τι για άλλα. Εμείς ε, ίσως θα θέλαμε και άλλες αλλαγές και για να πετύχουμε το στόχο μας ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση αυτών των ταμείων ας πούμε αλλαγή σε θέματα όσον αφορά τις, τους ελέγχους και μια καλύτερη διάφανη διαχείριση των ταμείων έτσι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το πεδίο όλο αυτό των ενεργειών και αλλά έχουμε μόνο μία δυνατότητα εδώ στην Επιτροπή σύμφωνα με τη δικασία να πούμε αν συμφωνούμε ή όχι με αυτή την αλλαγή του κανονισμού. Και εγώ νομίζω ότι κρατώντας υπευθυνή, τηρώντας υπευθυνή στάση, θα πρέπει να πούμε ότι συμφωνούμε. Εντάξει, θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα πράγματα και γι' αυτό εργαζόμαστε, όπως το είπε και η Επίτροπο, σε μια ομάδα εργασίας για να δούμε ως με δυνατότητες απλοποίησης και βελτίωσης αυτών των διατάξεων. Αλλά τώρα αυτό που χρειάζεται είναι να δώσουμε μια απάντηση σε αυτή την κατάσταση και θα πρέπει να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα και να μην βάλουμε εμπόδια στον ολοδρόμο και όλα αυτά θα πρέπει να περαιτωθούν όσο γίνεται συντομότερα να δείξουμε στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να δείξουν υπεύθυνη στάση να εφαρμόσουν όλα τα μέσα για να επιταχυνθεί η διαδικασία και θα δούμε και τη δυνατότητά μας πώς δηλαδή η Ευρώπη θα μπορούσε να βοηθήσει για να ξεφύγουμε από τη σημερινή οικονομική κρίση. Αυτά και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πέρες. Πολύ σημαντική έκθεση. Αλλά σήμερα θα κάνουμε μια πρώτη συζήτηση οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε και κάποιες συστάσεις γιατί τον Φεβρουάριο θα ξαναπαρουσιάσουμε αυτή την έκθεση και θα την ψηφίσουμε τον Μάρτιο. Οπότε, ποιος είχε ζητήσει τον λόγο, κυρία Γέλεβα. Ναι. Σας ευχαριστούμε. Εγώ από πλευράς ομάδας μου, σαν εισηγήτρια, θα ήθελα να επαναλάβω κατά κάποιο τρόπο τα όσα είπε η κυρία Περέζ και να πω ότι δεν πρόκειται βέβαια για την καλύτερη δυνατή διαδικασία, δεν μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγές, είτε συμφωνούμε είτε όχι. Και ακούσαμε και την κυρία Χίμπνερ που είπε ποια είναι η διάθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής να υπάρξει μια άμεση αντίδραση και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ως επιθυμούν γοργές λύσεις στην οικονομική αυτή κρίση. Εδώ λοιπόν εμείς θα πρέπει να πούμε ναι ή όχι στην πρόταση της Επιτροπής. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να δεχτούμε το ότι οι προτάσεις της Επιτροπής είναι αρκετά καλές, πάνε, οδηγούν προς την καλή, σωστή κατεύθυνση και έτσι να απαντήσουμε όσο γίνεται συντομότερα και με την πολιτική συνοχής ε, να προσφέρουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ενεργήσουν σωστά και αυτές οι προτάσεις αποσκοπούν στο να απλοποιήσουν την όλη διαδικασία και να επιταχύνουμε την διάθεση των κονδυλίων με όλα τα όργανα τα οποία θα πρέπει να συμμετάσχουν και μάλιστα εξ ονόματος της πολιτικής συνοχής. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό το δρόμο, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό και να μην ξεχνάμε ότι οι προτάσεις αυτές έχουν να κάνουν με το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης και εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Στήλερ κατόπιν ζήτησε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια και την προηγούμενη ομιλήτρια για τα σχόλια της. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί βεβαίως ε, μας απογοητεύεται ότι δεν έχουμε χρόνο, ο χρόνος δεν υπάρχει αλλά όταν μιλάμε με τους ανθρώπους επιτόπου για τα διαρθρωτικά ταμεία, ένα από αυτά τα οποία μιλάνε είναι βεβαίως η ε, παρέμβαση. Είναι ωστόσο ένα παράδειγμα, π.χ. το 45% των χρημάτων προέρχεται από την Ευρώπη που πρέπει βεβαίως να συμπληρωθεί από ένα 55% από το κράτος μέλος. Το να αλλάξει αυτό και να γίνει 55% ευρωπαϊκά κοντήλια και 45% από το κράτος μέλος είναι η διαφορά από το να είναι κάτι απλά δυνατό με το να γίνει κιόλα. Θεωρείτε λοιπόν πως οι αλλαγές ε, στα διευθυντικά ταμεία βοηθούν ε, θα κάνουν αυτή την διαφορά, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Γνωρίζω μιλώντας με μικρές επιχειρήσεις πως είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθούν κάποια κονδύλια για να προχωρήσουν κάποιες συμπράξεις που θα δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας και τα λοιπά. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσουν η αν εάν θεωρεί πως ε, όσον αφορά τη συγκεκριμένη πτυχή θα βοηθήσει αυτή η πρόταση. Αυτό και είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι εντάξει βρισκόμαστε μεταξύ σκύλας και χάριτης και σας ευχαριστώ για τη δουλειά την οποία κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάλμα. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.